Οκτωβρίου επαλήθευσε την εντολή του κυρίου Γιασένκο Σελιμούβιτς και την επικύρωσε με ισχύ από 30, 30 Σεπτεμβρίου 2015. Υπάρχουν αντιρρήσεις προς την εντολή αυτή. Εγκρίνεται λοιπόν.